Θα πρέπει, ε, πρόσφατα επίσης η Κομισιόν ε, εξήγησε τις λεπτομέρειες αυτής της διαδικασίας. Ευχαριστούμε πολύ. Κλείνει η συζήτηση. Αύριο, ε, Τρίτη, 8 Οκτωβρίου στις 12 είναι η ψηφοφορία. Περνάμε τώρα στην έκθεση Έλλης. Δίνω το λόγο στον κύριο James Έλλης. Σε President, buonasera. colleagues, uh, good Καλησπέρα συνάδελφοι. Έχω τη χαρά να σας παρουσιάσω αυτή την έκθεση πρωτοβουλία από την Επιτροπή Προπολογισμών και ευχαριστώ τους συναδέλφου στην Επιτροπή που μου έδωσαν αυτή τη δυνατότητα. Ε, ο στόχος ε, είναι να δούμε που έχουμε φτάσει και τι μπορεί να γίνει ακόμα έτσι ώστε να υπάρχει αυτό το διοργανικό σύστημα για μακροπρόθεσμε τάσει. Υπάρχει σήμερα αλλαγή του παγκόσμιου συστήματος και ο στόχος είναι οι κοινοτικοί θεσμοί να μπορούν να έχουν τα μέσα να λαμβάνουν υπόψη τους μακροπρόθεσμες τάσεις οποτεδήποτε λαμβάνουν επίκαιρες αποφάσεις. Η ε, κοινοτική πολιτική θα εξαρτάται όλο και περισσότερο από τον έγκαιρο εντοπισμό αυτών των μακροπρόθεσμων τάσεων που επηρεάζουν τις ε, επιλογές της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει όμως να αυταπατώ ότι ο στόχος είναι να ξέρουμε τι θα συμβεί στο μέλλον. Στην ιστορία υπάρχουν πάρα πολλοί ε, που πίστευαν ότι μπορούσαν να ε, προβλέψουν τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Το 62 παραδείγματος χάρη ήταν ε, τότε οι Beatles και πολλοί πίστευαν όμως ότι η μουσική pop δεν θα είχαν κανένα μέλλον. Λάθος βέβαια. Επίσης ε, το 2008 ε, κανείς δεν πίστευε ότι θα στερεωθούν, θα ενισχυθούν τόσο πολύ το Google και το Facebook. Εμείς προτείνουμε ότι θα πρέπει να μπορεί κανείς ε, να προβλέψει ε, μια ανάλυση υψηλής ποιότητας έτσι ώστε οι πολιτικοί να το κάνουν αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα χρονικά διαστήματα. Μέχρι τώρα τι έχουμε καταφέρει. Το πρόγραμμα βασίζεται σε δύο γραμμές του προεπολογισμού. Το πιλωτικό πρόγραμμα ε, οδήγησε σε ένα έγγραφο για τις παγκόσμιες τάσεις ε, μέχρι το 2030 σε έναν περίπλοκο κόσμο υπό την ε, αιγίδα του ΑΣΕ στο Παρίσι επισημένονται τρία βασικά θέματα. Το πρώτο είναι ε, το ότι το άτομο αποκτά όλο και περισσότερες δυνατότητες λόγω της τεχνολογικής αλλαγής. Δεύτερον, ε, βελτιώνεται ε, και αυξάνεται η ε, μεσαία τάξη, μειώνεται η φτώχεια και τρίτον προκύπτει ένας πολυπολικός κόσμος όπου ε, μη κρατικοί φορείς παίρνουν όλο και μεγαλύτερο ρόλο. Σε δεύτερη λοιπόν φάση αποδίδεται μεγαλύτερη σημασία σε οικονομικές και άλλες τάσεις και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να εντοπίσουμε εκείνες τις τάσεις που θα επηρεάσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά επόμενα πέντε χρόνια. Φτάνουμε στο 2014 και νομίζω ότι μπορεί να γίνει μια μεγάλη συζήτηση για τις αναδιόμενες απόψεις. Ένα έγγραφο εργασία θα σας κατατεθεί σύντομα με απόψεις που θα έχουν συγκεντρωθεί από όλες αυτές τις πηγές πριν ολοκληρώσουμε στο έγγραφό μας το τελικό ε, κατά τα μέσα του επόμενου έτους. Παράλληλα στο μέλλον, δηλαδή τους επόμενους μήνες, ε, παράλληλα με αυτή την έκθεση θα επεξεργαστούμε και την διοικητική συνεργασία, μια διοργανική συμφωνία όπου κάθε εταίρος θα συμφωνήσει να συμμετάσχει ε, στη συμφωνία. Επιπλέον η διαδικασία στη διαδικασία προβλέπεται και ένα συστότοπος, έτσι ώστε ε, να λαμβάνονται υπόψη οι παγκόσμιες τάσεις. Από τη στιγμή που θα υπάρχει αυτό το σύστημα θα μπορεί να προσφέρει τα απαραίτητα στοιχεία στις ε, ε, αρχές του προϋπολογισμού ή ε, γενικά ε, θα προσφέρονται άλλα στοιχεία για τις παγκόσμιες τάσεις. Έτσι λοιπόν, χάρη της δουλειάς πάρα πολλών οργανισμών, ε, το πρόγραμμα έχει ως στόχο να επιτύχει το στόχο του και το σχεδιασμό του. Εάν τα καταφέρει, θα προσφέρει αξιόπιστα έγγραφα, τα οποία θα βοηθούν να προετοιμάζουμε τις αποφάσεις με διαφανή τρόπο. Κατά το παρελθόν, πολλοί έλεγαν ότι υπερισχύει ο ισχυρός. Στον αυριανό κόσμο, όσοι είναι καλύτερα ενημερωμένοι, αυτοί κατά πάσα πιθανότητα θα επιβιώσουν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στη διαδικασία Catch the Eye, το λόγο έχει ο κύριος Πλένκοβιτς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είμαι μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τέος διπλωμάτης ο οποίος έχει περάσει μεγαλύτερο μέρος της ζωής του σε τμήμα σχεδιασμού. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Έλλης για την εξαίρετη εκθεσή του. η οποία έχει να κάνει με τη στρατηγική ανάλυση. Πρόκειται για τη διοργανική συνεργασία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Πιστεύω ότι όταν πρόκειται για την οικονομία, για την ε, παγκόσμια διακυβέρνηση, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας διάφορα στοιχεία για να σχεδιάσουμε το μέλλον μας. Γιατί έτσι θα χρησιμοποιήσουμε με πιο κατάλληλο τρόπο τα κονδυλιά μας. Για την πολιτική συνοχής, για παράδειγμα, έτσι θα μπορέσουμε να πετύχουμε καλύτερα τους στόχους που νοιάζουν τους πολίτες. Πιστεύω λοιπόν ότι έτσι μπορούμε να είμαστε πιο υπεύθυνοι. Γι' αυτό συστήνω το κείμενο αυτό και ελπίζω να τεθεί σε εφαρμογή και να χρησιμεύσει για την περίοδο 2012-2014. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, η κυρία Δαμανάκη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Έλλης, για την ομιλία του, για τόσα είπε, αλλά και για το έργο του όσον αφορά την έκθεση αυτή. Και να τον ευχαριστήσω επίσης για την Προεδρία που είχε αναλάβει στην Task Force για, την, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Στρατηγικής και Πολιτικής Ανάλυσης. Πρόκειται για ένα διοργανικό σχέδιο που είναι πολύ σημαντικό για μας. Θέλω επίσης να το συγχαρώ για την πρωτοβουλία που ανέλαβε προκειμένου να εφαρμοστεί το σύστημα αυτό πολιτικής και σε επίπεδο δοκιμαστική δράσης αλλά και προπαρασκευαστικής τώρα Πράγματι, ο κόσμος αλλάζει με μεγάλη ταχύτητα. Το αποτέλεσμα είναι ότι όσοι αποφασίζουν για την πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση μερικές φορές δυσκολεύονται να προλάβουν τα γεγονότα. Αυτό το σύστημα πολιτικής πάντως προσπαθεί να δει πώς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορούν να συνεργαστούν καλύτερα για να εντοπίσουν τις παγκόσμιες τάσεις, να τις αναλύσουν καλύτερα και να δουν τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν αυτές, άρα και τι πολιτικές απαντήσεις πρέπει να δώσουμε. Συνεπώς, πρόκειται για ένα πραγματικά μοναδικό διοργανικό σύστημα όπου συμμετέχουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης με στόχο την ανάλυση των ε, παγκοσμίων τάσεων και της ε, γενικότερης παγκόσμιας διακυβέρνησης. Του χρόνου αυτή, αυτό το σύστημα το Ευρωπαϊκό Στρατηγικής και Πολιτικής Ανάλυσης θα ετοιμάσει έκθεση προς τους πρόεδρους των θεσμικών οργάνων προκειμένου να γίνει ανάλυση μέσα στον επόμενο κύκλο. Η διοργανική Task Force εξετάζει επί του παρόντος τι μορφή και τι μόνιμο σύστημα τελικά πρέπει να εφαρμόσουμε. Οι εργασίες συνεχίζονται και ελπίζουμε ότι έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ξέρετε ότι θα συνεχίσει να συνεισφέρει θετικά στις συζητήσεις αυτές. Εύχομαι λοιπόν ότι καλύτερο στον εισηγητή και πρόεδρο της ε, Ομάδας Εργασίας για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Στρατηγικής και Πολιτικής Ανάλυσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Έληξε η συζήτηση για αυτό το θέμα. Αύριο στις 12 το μεσημέρι θα γίνει η ψηφοφορία. Και τώρα περνάμε στο επόμενο θέμα που είναι η έκθεση Ρέγνερ. Το λόγο έχει η κυρία Εβελίν Ρέγνερ, παρακαλώ.